θα υπενθυμίσω ότι από τα έξι μέλη της Εθνικής Διεύθυνσης, τα πέντε είναι κατά του καθεστώτος και το ίδιο ισχύει και για όλα τα μέλη της Επαναστατικής Συνόδου της κυβέρνησης του 1977, όπως και χιλιάδες σύντροφοι σαντινίστας. Είναι αυτοί οι πραγματικοί σαντινίστας που σήμερα διώκονται από τον Τελή Ορτέγα επειδή υπερασπίζουν όσα είχε υπερασπίσει και αυτός κατά τους ομόσα την ελευθερία και την αξιοπρέπεια καταστολή, εκατοντάδες νεκροί, διαφθορά, παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η Νικαράγουα του Ορτέγα και ε, δυστυχώς το υπερασπίζουν μόνο ε, επαναστάτες του Σαλονιού γιατί αυτούς δεν τους ενδιαφέρει η Νικαράγουα αλλά η δική τους ιστορία, η μακρινή επανάσταση, άλλη επανάσταση και όχι δική τους. Το ψήφισμα που θα έχουμε αύριο αποτελεί αποτέλεσμα συνολικής ε, συμφωνίας. Ε, τίθεται ε, το θέμα της επιβολής προσωπικών κυρώσεων στον Ορτέγα και της κυβέρνησης που καταστέλει και φυλακίζει τους δικούς του συντρόφους και τον ίδιο του το λαό. Και εγώ από την ψυχή μου θα πω αυτό που είπα και το 77. Ζήτω η ελεύθερη Νικαράγουα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πιμέντα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα κάποιες από τις παρεμβάσεις και πολλές φορές αναρωτιέμαι αν μιλάμε για την καταστολή και για τους φυλακισμένους στη Γαλλία και στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο ε, ουσιαστικά ε, τρέφει τη στρατηγική Τραμπ. Ε, ξέρετε ότι η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης ήθελε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος και να αποφύγει τις νοφιλελεύθερες συνταγές του Δουνουτού. Ξέρετε ότι ε, υπήρξε, υπήρξαν αντιδραστικοί τομείς της δεξιάς που προκάλεσαν νεκρούς ε, και βίες συγκρούσεις. Αυτή η βία ε, δεν ήταν κατά της κυβέρνησης μόνο αλλά και κατά μελών του μετόπου Σαντινίστε. Με αυτή τη πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει έναν ευρύ διάλογο προσπαθούν να βρουν ειρηνικές λύσεις. Η κυβέρνηση τον ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις και απειλεί την Ικαράγουα με οικονομικό βέτο και ε, παραβιάζει το χάρτη ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Χρησιμοποιείται αυτός ο τρόπος για να επιτεθούν σε ορισμένους λαούς όπως στην Ικαράγουα η οποία πρέπει να έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και θα πρέπει να καθορίσει το δικό της κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό δρόμο. Κύριε Πιμέντα, έχετε μία μπλε κάρτα από την κυρία Γκόμες. Όχι, κύριο Σκοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ιστορία δεν μας διδάσκει τίποτα από ό,τι φαίνεται, κυρίως στην περίπτωση του Ικαράγουα το 1970. τη δεκαετία του 70 είχε θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του έναντι τη δικτατορία. Ο Ντανιέλ Ορτέγα τώρα, ο Ορτέγα δεν έχει ένα δικτάτορα να πολεμήσει. Τώρα αυτός έχει γίνει δικτάτορας η χώρα. Ε, βρίσκεται όμως ε, σε μια κατάσταση όπου βλέπουμε λογοκρισία, βασανιστήρια, εξαφανίσεις για να μην μιλήσουμε για σταγματικές ε, τροποποιήσεις που έχουν επιτρέψει στον Ορτέγα ε, να αδράξει τις ελευθερίες. Ε, δεν ενδιαφέρει όμως τον κόσμο αυτή η δικτατορία γιατί η Νικαράγου είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες ε, του πλανήτη και δεν βασίζεται στην υποστήριξη του λαού αλλά σε όσους πυροβολούν το λαό. Και θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να έχουμε ατομικές κυρώσεις που θα επιβληθούν ε, κατά των υπεύθυνων του καθεστώτος που ε, προβαίνουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το έγγραφο που συζητάμε περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία με τα οποία συμφωνούμε για μια χώρα διαιρεμένη που από ό,τι πολλοί λένε θα είναι η επόμενη Βενεζουέλα. Όμως ε, υπάρχει μια παράληψη. Δεν γίνεται λόγος για κάτι που όλοι γνωρίζουν. Ξέρει η διεθνή κοινή γνώμη ότι σχεδόν πάντα, πάντοτε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήθελε να γνωρίσει ότι αυτό το καθεστώς έχει φιλοξενήσει για δεκαετίες ε, τους χειρότερους ε, τρομοκράτες μεταξύ των οποίων μέλη των ερυθρών ταξιαρχιών. Υπάρχει μια έκκληση που προέρχεται από τον τελευταίο πρόεδρο της Επιτροπής ε, Μόρο να επιστρέψει τελικά ε, στην Ιταλία μετά από τόσες πιέσεις, ένας από τους πιο επικίνδυνους ε, από το πιο επικίνδυνα μέλη των ερυθρών ταξιρχιών που δεν έχει περάσει ούτε καν μια μέρα στη φυλακή. Ο Διέσο Κασιμίρη, ο οποίος μια χαρά τα περνάει και βρίσκεται στη Μανάγουα. Δεν μιλάτε για το σκάνδαλο αυτό. Ίσως γιατί για πολύ καιρό ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε δώσει την ίδια Αλλά ίσως ε, θα ήταν τώρα καιρός να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εμείς ε, ζητάμε η Ευρώπη να ζητήσει την άμεση έκδοση στην Ιταλία αυτού του εγκληματία, αυτού του δολοφόνου. Είναι στιγμή να ξυπνήσει επιτέλους η Ευρώπη και να μην υπάρχει πλέον ομερτά απέναντι σε αυτούς τους τρομοκράτες. Ποτέ δεν ασχοληθήκατε με αυτούς. Δεν σας ενδιαφέρουν τα θύματα της ε, τρομοκρατίας της Ιταλίας, όμως τα θύματα ζητούν επιτέλους δικαιοσύνη και αυτό είναι ντροπή. Θα πρέπει να επανορθώσετε αμέσως αυτή την πολύ σοβαρή παράληψη απέναντι στη διεθνή κοινή γνώμη και στα θύματα της τρομοκρατίας και των ε, δολοφόνων του Πρόεδρου Μόρου. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, βοηθήστε μας, παρακαλώ. Αυτό ε, ακούστηκε από τις φυλακές, από τους κρατούμενους που καθημερινά ξυλοκοπούνται, στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και δεν τους ε, επιτρέπουν να δουν ε, τις οικογένειές τους. Είναι αθώοι. Στην φυλακή βρίσκονται απλώ έχουν, επειδή υπεράσπισαν τις ιδέες τους σε μια χώρα που κυβερνάται από ένα τύρανο που δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία, ούτε γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε υπάρχει ελευθερία έκφρασης και το συνέχιστε οι γυναίκες ε, δεν παραδίδονται και μας το ομολόγησαν με πραγματική δύναμη. Βάσει όλων όσων μας είπαν και βάσει όσων είδαμε, απαιτούμε από τις ε, αρχές των φυλακών ε, και τον Αντιπρόεδρο αλλά και τον Ρωτέγκα να μην υπάρχουν αντίπεινα. Μάλιστα, ο Τύρανος το αντίθετο έκανε και συνέχισε να αυξάνει την καταστολή μέχρι τώρα, 1,5 μήνα μετά, να φτάσουμε σε μια αβίωτη κατάσταση. Η πραγματικότητα της Νικαράγουας είναι ιδιαίτερα ενισχυτική τουλάχιστον ε, για όλους όσους αισθανόμαστε δημοκράτες και επερασπίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους πολίτες οποιασδήποτε χώρας. Από τότε που ξέσπασε η κρίση στην Ικαράγουα, έχουμε πάνω από 300 νεκρούς, πάνω από 1.400 τραυματίες, περίπου 700 πολιτικούς κρατουμένους και περίπου 50.000 εξόριστους. Δεν σας φαίνονται ε, πολύ ψηλά αυτά τα νούμερα. Εμένα μου φαίνονται ανατριχιαστικά. Και θεωρώ ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορο ούτε μια στιγμή ακόμη. Πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη, πρέπει να δράσει. Κύριε Επίτροπε. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ικαράγουα αποτελεί μέρος της ευθύνης της δικής σας επιτροπής. Η Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί και να δείξει την ισχύ της. Ένα καθεστώ όπω το Ορτέγα Μουρίγιο δεν μπορεί να ζητά διάλογο με την αντιπολίτευση. Είναι φάρσα αυτό. Για να υπάρξει πραγματικό διάλογο, χρειάζεται η άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και η πάυση κάθε μορφή κακοποίηση ή καταστολή του λαού. Φτάνει πια η Νικαράγουα αξίζει να ζήσει ειρηνικά και οι ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου θα έπρεπε ομόφωνα να στείλουν ε, αυτό το μήνυμα στον επεναστάτη που πρόδωσε μια χώρα. Αυτοί οι τύρανοι που έφτασαν με ψευδοδημοκρατικά τεχνάσματα για να παρουσιάσουν ε, κάποια δημοκρατικά διαπιστευτήρια φοβούνται τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας και επίσης φοβούνται πως χάσουν τα προνόμια ε, που έχουν κατακτήσει. Εδώ υπερασπίζω λοιπόν την επιβολή κυρώσεων κατά το μελών της κυβέρνησης Ορτέγα, αν ε, δεν σέβονται την αρχή του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και τις ελάχιστες αρχές ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η δημοκρατική ρήτρα ώστε η Νικαράγουα να αποκλειστεί από τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Αμερική. Ευχαριστούμε. Κυρία Βαλενσιάνο. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, αν και λείψα, θέλω να πω στον συνάδελφο που εμένει να πέσω ότι στην Ισπανία δεν έχουμε πολιτικούς κρατουμένους. Η Ισπανία είναι ένα κράτος δικαίου μια σύγχρονη και παγιωμένη δημοκρατία και όσες φορές και να το λέτε δεν θα δεχτούμε να λέτε ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Ελπίζω κάποιο να του στείλει το μήνυμα παρότι λείπει. Δεύτερον, πολλοί λίγοι στον προοδευτικό κόσμο συζητούν ότι ο Ντενίλ Ορκτέγα έκανε ε, κάτι πολύ φαύλο ε, εξ ονόματος μιας ε, επανάστασης που εξέπληξε όλο τον κόσμο και θαύμασε όλος ο κόσμος. Ε, όμως βάσει αυτής της επανάστασης ε, τελικά οικοδόμησε ένα αυταρχικό καθεστώς. Γι' αυτό αποφάσισε το Κοινοβούλιο να δράσει και γι' αυτό μια, μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου με επικεφαλή στον κύριο Χαουρέγη αποφάσισε ότι θα έπρεπε να υψώσουμε τη φωνή μας στο Κοινοβούλιο για να την ενώσουμε με τη φωνή του συνόλου της δημοκρατικής αντιπολίτευσης του λαού της Νικαράγουας για να ζητήσουμε ένα διάλογο, αλλά μόνο όταν ε, πληρωθούν οι ελάχιστοι όροι, οι ελάχιστες προϋποθέσεις. Ελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, ελευθερία έκφρασης και να σταματήσει η καταστολή. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, ενώ συνεχίζεται η καταστολή. Αυτή είναι η φωνή του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να την ακούσει το καθεστώ Ορτέγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλενσιάνο. Ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Uh, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ξεκίνησαν ε, οι διαδηλώσει στην Καράγουα το 2018 ήταν ε, εμφανές ότι δεν ήταν διαδηλώσει κατά των μέτρων λιτότητας, αλλά ε, Διαμαρτυρίε των ανθρώπων που ήθελαν να αγωνιστούν για τα δικαιώματα και τι ελευθερίε του. Και ήταν ε, ένας αγώνας ε, για την δημοκρατία σε μια απολωμένη χώρα. Από τότε εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάνω από 700 φυλακίστηκαν, κυρίως με βάση πολιτική λόγους και η κυβέρνηση διασφάλισε ότι δεν θα γίνουν αντίπεινα κατά τους ακτιβιστές. Αυτό αντανακλάται και στο ψηφισμά μας. Ε, βλέπουμε, ε, θέλουμε να ε, ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με ελπίδα και δυστυχώς σταμάτησαν. Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρέχει μια λύση στην κρίση αυτή. Είναι ο λαό τη Νικαράγουα που θα πρέπει να δουλέψει μαζί για να απειλήσει τη διαφορά. εμεί θα δουλέψουμε για την προάσπιση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπά. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Πίτροπε. Η καταστολή που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νακαράγουας, η απέλαση των ε, μαρτύρων που δεν βολεύουν ε, είναι μια στεπτική για να εμποδίσει την πολιτοίτευση. Ε, σήμερα εφαρμόζονται οι μέθοδοι του ΣΟΜΟΣ, αυτό που είχαν καταπολεμήσει οι ίδιοι. Το, ε, μας το είπαν μέλη της Επιτροπής που επισκέφθηκαν τη χώρα τον Ιανουάριο. Μια βιώσιμη έξοδος από την κρίση απαιτεί το τέλος της καταστολής και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, αποτελεί το τέλος της παρενόχλησης. Πρέπει να αποκατασταθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος. Όπω αναφέρει και το κοινό ψήφισμα, η εξωτερική υπηρεσία τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει σταδιακά κυρώσει ε, χωρί να θυγεί ο λαό, αλλά να ποινικοποιούνται τα μέλη τις κυβέρνησεις που μπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να επικαλεστούμε την δημοκρατική ρήτρα για να μπορέσουμε να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις με την Ικαράγουα. Ευχαριστώ, κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, ήμουνα στην Ικαράγουα τέλη Ιανουαρίου που είδα στην ε, φυλακή των γυναικών την Αμαγιά Κοπένς, ε, φοιτήτρια ιατρικής, 23 ετών. Ε, ήταν στο κίνημα και κρατείται για πολιτικούς σκοπούς. Η Αμαγιά και οι συντρόφισσες της σταμάτησαν την απεργία πείνας και είμαι πολύ ανήσυχη για τις συνθήκες υγιεινής κράτησής τους. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να υποφελούνται ε, παρακολούθησης, ιατρικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τους ελάχιστους κανόνες του 1955 για τη μεταχείριση των κρατουμένων των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσφατα, μια 100 κρατούμενοι φυλακίστηκαν σε εισαγωγικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι υποκατοίκον περιορισμό υπό συνεχή επιτήρηση. Ε, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε την ε, ε, διεθνή γνώμη για την κατάσταση των κατουμένων που είναι 670. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας. Ο κύριος Μηγιάννη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από ένα μήνα, σε αυτό το ημικύκλιο, όπως είπε και ο κύριος Μάτο, καταγγείλαμε την περίπτωση κάποιων γυναικών που είχαν φυλακιστεί στην φυλακή Εσπεράνσα, Ελπίδα, και ήταν αντικείμενο ε, ουσιαστικά αντιπίνων επειδή μίλησαν με τους ευρωβουλευτές. Ε, θα πρέπει να σταματήσει η στέρηση της ελευθερίας αυτών των νέων και των λοιπόν πολιτικών κρατουμένων καθεστώς Ορτέγα θα πρέπει να λάβει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις ε, με την αντιπολίτευση της Αστικής Συμμαχίας ε, και να σεβαστεί την ε, το αίτημά του στην απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, όπως και άλλους όρους που θέτουμε στο ψήφισμα. Από πέρσι έχουμε περίπου 400 νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες ξεκίνησε η κρίση αυτή από τις διαδηλώσεις ε, κατά του καθεστώτος. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση για την επίλυση της κρίσης. Βάσει του ψηφίσματός μα, ε, του περσινού Μαΐου θα πρέπει να έχουμε δίκαιες και αξιοπιστέ εκλογέ. Είναι απαραίτητο γι' αυτό να υπάρχει εκλογική μεταρρύθμιση συμπεφωνημένη. Εγώ θέλω να ζητήσω από ε, τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω από την Υπηρεσία εξωτερική δράση ε, να παρακολουθεί του σύνεγγες τη εξέλιξη στην Καράγουα. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να επιβληθούν ειδικέ κυρώσεις κατά των υπευθύνων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε την ε, ε, αποπομπή της ε, Νικαράγουας από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Δηλαδή, να ενεργοποιήσουμε τη δημοκρατική ρήτρα της Συμφωνίας. Και επίσης, και για τους πολίτες Νικαράγουας και της Βενεζουέλας εύχομαι ελευθερία, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και ευημερία. Και πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό από αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Γκόμες. Πρόεδρε. 20 χρόνια, τα πρώτα 20 χρόνια τα πέρασα σε δικτατορία. Γι' αυτό αναγνωρίζω μία όταν τη βλέπω και αυτό είδαμε στην Καράγω το 2011 και το περασμένο Ιανουάριο. Μάλιστα υπήρχε μεγαλύτερη διαφθορά και εκδίκηση κατά του λαού από τους ε, δρόμους όπου είχαμε ε, περιπολίες του στρατού και της αστυνομία ε, μέχρι τις φυλακές όπου τόσοι να είχαν φυλακιστεί και τους ε, μεταχειρίζονταν ως τρομοκράτες. Λούσιο Πιγέρα, Ιλάντα Χερές, Μιγέλ Μόρα, Ελέσια Μουνιός και τόσοι άλλοι Ακόμη και η Μάγια Κοπένς που με τους συντρόφους της από τις 27 Φεβρουαρίου είναι σε απεργία πείνας. Πολλοί στην Ικαράγουα μας είπαν ότι οι Ορτέγα δεν θέλουν να διαπραγματευτούν, θέλουν να κερδίσουν χρόνο μέχρι να δουν τι θα γίνει στη Βενεσουέλα. Αυτό επαληθεύτηκε κύριε Επίτροπε με την πρόσφατη προσπάθεια διαπραγμάτευσης και δεν ε, πέτυχαν τίποτα, ούτε καν την απελευθέρωση των 100 κρατουμένων. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει τη διαφορά στην Καραγουά, να συνεργοποιήσουμε την, την ε, δημοκρατική ρήτρα και πρέπει να επιβάλλουμε συγκεκριμένες κυρώσεις ε, απέναντι, μάλλον επί των υπευθύνων και στους Ορτέγα και Μουρίγιο και να απαγορεύσουμε και τις θεωρήσεις. Η Ορτέγα Μουρίγιο και όσοι τις υποστηρίζουν θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην εθνική ή διεθνή δικαιοσύνη προκειμένου να αλλάξει κάτι στο κέντρο εξουσίας στη Μεράγουα. Ο κύριος Φαριά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, είμαι Πορτογάλος αλλά θα μιλήσω ισπανικά γιατί θέλω να απευθυνθώ σε πολλούς φίλους από την Ικαράγουα και σε όλους ε, τους αντιπολιτευόμενους οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται για την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελευθερίας στη χώρα τους και να απευθύνομαι σε όλους εσάς, κυρίως στους γονείς που βλέπετε τα παιδιά σας να δολοφονούνται από παραστριωτικού και την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σε όλους τους φοιτητέ ε, που ε, διακυβεύουν ε, τη σταδιοδρομία τους και το μέλλον τους λόγω της ειρηνικής συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις και σε όλους αυτούς τους θαραλέου ανθρώπους οι οποίοι συνελήφθησαν επειδή απλώς ήθελαν να εκφράσουν την άποψή τους. Πολλοί φυλακισμένοι ε, σε απάνθρωπα κελιά που ε, δεν αξίζουν ούτε για γουρούνια. Έχουμε την Λούσια ε, Μπουλμπάου που ε, θέλω να τη χαιρετήσω από εδώ. Αυτό ήταν το σενάριο που μπορέσαμε να δούμε και επιβεβαιώνουμε ότι το πραξικόπημα που ενορχιστρώνεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες ήταν απλώς προπαγάνδα ε, του καθεστώτος Ορτέγα Μουρίγιο μετά από την ε, επίσκεψή μας εντατικοποιήθηκε η καταστολή και ο κύριος Ορτέγα πρέπει να δείξει ότι δεν χρησιμοποιεί τον ενθετικό διάλογο ως μανούβρα για να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αποδεικνύεται μόνο με το τέλος της καταστολής ε, και ε, να ακυρώσει τις δίκες των κρατουμένων. Ε, επίσης, θα πρέπει να ε, δώσει πίσω τα περιουσιακά στοιχεία που έχει δημεύσει και να επιτρέψει οι εθνικές και δημοτικές εκλογές να γίνουν νωρίτερα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει συγκεκριμένες και ατομικές κυρώσεις στους υπεύθυνους κυβέρνησης της ε, Νικαράγος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να ενεργοποιηθεί η δημοκρατική ρήτρα της συμφωνίας. Όπως λέγεται στη χώρα μου, δεν μπορούμε να κλείσουμε ε, μία πόρτα αφήνοντας ανοιχτό ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο που μπορεί να σημαίνει στην περίπτωση αυτή ότι εκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων φορολογουμένων μπορεί να χρηματοδοτήσουν ένα ε, καθεστώς που ήδη έχει προκαλέσει πάνω από 300 ε, νεκρούς, 1.000 τραυματίες και χιλιάδες εξόριστους. Κύριε Ζωρίνιο, η δημοκρατία δεν είναι μοντέλο ε, ανεξάρτητο από τους λαούς. Σε... Χρειάζονται κάποιοι όροι για να υπάρξει δημοκρατικό καθεστώς. Ε, αυτές τις αξίες εμείς υποστηρίζουμε στο δικό μας πρόγραμμα και γι' αυτό εμείς ε, θέλουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές και παγκοσμίω. Είναι αρχές που βασίζονται στο κράτος δικαίου και στην αξιοπρέπεια του λαού. Με αυτές τις αρχές ε, ουσιαστικά προσπαθούμε να ε, δώσουμε και στο λαό της Βενεζουέλας τη δυνατότητα να ζει ελεύθερος και Επίσης, ε, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το αυταρχικό καθεστώ τη Νικαράγουα. Έχουμε μηχανισμού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που μα προσφέρει το διεθνέ δίκαιο, για να τοποθετούμε δίπλα στο λαό τη Νικαράγουα για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια των λαών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε με θάρρο Και το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε αύριο σε αυτόν τον οίκο αποτελεί τη σχετική απόδειξη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κύριο Σωσή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ ανήκω σε μία γενιά που στην ε, εφηβεία της παρακολούθησε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ελπίδα τη Σανδινιστική Επανάσταση στην Καράγουα. Μάλιστα, θυμάμαι ότι κάθε μέρα περιμέναμε ειδήσει ε, που να προέρχονται από αυτή τη χώρα και θυμάμαι και τι ε, μέρες που γιορτάσαμε με μεγάλη χαρά την πτώση του δικτάτορα Σομόσα και τη νίκη των ε, ε, Και όμως παρόλα αυτά αυτό το καθεστώς απέτυχε απέναντι στο λαό του. Δεν ε, ήταν στο ύψος των ιστορικών του ευθυνών. Και τώρα υπάρχει παραπληροφόρηση εφευρίσκει εξωτερικούς εχθρούς για να καλύψει τα δικά, τις δικές του αποτυχίες Σύμφωνα και με το καθεστώς των Πολυβεριανών στη Βενεζουέλα, έχει προδώσει ε, το καθεστώς ε, του Ορτέγα τις δημοκρατικές ε, αξίες, καταστέλει τις δημοκρατικές ελευθερίες. Όμως εξ ονόματος αυτών των δημοκρατικών ελευθεριών εμείς θα πρέπει να καταγγείλουμε κάθετα αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Καραγό και αυτό το ψήφισμα αυτό ακριβώς κάνει. Αναφέρουμε ε, τις ε, παραβιάσεις ε, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμε να αποπομπεί η Νικαράγου από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής και αυτό στο όνομα μιας λέξης δημοκρατίας. Στο όνομα αυτής της λέξης έγινε με δημοκρατική επανάσταση και μπορούμε να πούμε σήμερα δυστυχώς ότι προδόθηκε τα τελευταία χρόνια η επανάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο ΚΑΤΣΔΙ. Η κυρία Σόντρουβα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους που ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση και που πρότειναν ε, την γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα αλλά και άλλους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, διότι αυτό που συμβαίνει στην Ικαράγουα αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Η κατάσταση είναι πολύ παρόμοια με αυτή της Βενεζουέλας και της Κούβας. Ε, ένα ελεκιστικό κατεστώς υπό τον ε, Ορτέγα που ξεκινάει από τον ψυχρό πόλεμο μετά ε, και βρίσκεται για δεκαετίες στην ηγεσία. Έχει διευθύνει τη χώρα, χειραγωγεί τις εκλογές, δεν αφήνει τη χώρα να λειτουργήσει, δεν αφήνει τις εκλογές να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποφυλακιστούν 700 κρατούμενοι είναι υποκράτηση, ε, ε, υποβασανιστήρια, διώκονται μαζί με δεκάδες άλλους διαδηλωτές που διαδηλώνουν κατά το πολέμου. Ήρθε η στιγμή το Ευρωκοινοβούλιο να υψώσει τη φωνή του κατά αυτής ε, της κατάστασης και της καταστολής που επικρατεί στην Εκαράγουα. Η αντιπολίτευση πρέπει να ξέρει ότι έχει την στήριξη όλου του πολιτικού φάσματος στην Ευρώπη. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπε ο συνάλφος εδώ πέρα ότι κοιτούσε τον Ορτέγα με ελπίδα όταν ήταν νέος. Εγώ ζούσα στην Τσεχοσλοβακία και θυμάμαι που ήρθε στην Τσεχοσλοβακία και αγκάλιαζε εκεί πέρα τους κομμουνιστές κυβερνώντες και τον πρόεδρο. Οπότε δεν προξενεί έκπληξη το τι έκανε τελικά. Είμαι πολύ επιφυλακτικός ε, κύριε Επίτροπε για τη δυνατότητα διαλόγου με τον Ορτέγα. Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι δημοκρατικές εκλογές και η εγκατάλειψη αυτού του πολιτικού δεινόσαυρου ανήκει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις για να γίνουν ελεύθερες εκλογές στην Καραγουά. Σας ευχαριστώ κύριος Νίμιτσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές ε, για το ότι θέλετε να βοηθήσουμε τον λαό της Νικαράγουας να βγει από την κρίση αυτή με τρόπο ειρηνικό. Η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου αυτού και της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ήταν πραγματικά υποδειγματική για να ακουστεί η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νικαράγουα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, για την προσωπική του προσήλωση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Νικαράκουα. Ακούσαμε προσεκτικά τους διάφορους βουλευτές ε, που επιθυναν έκκληση να ε, επιβάλλουμε κυρώσεις στην Νικαράγουα. Είμαι πεπισμένος πως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο θα παρακολουθήσουν την διαδικασία ενός πολιτικού διαλόγου που διεξάγεται, ελπίζουμε ότι θα διεξαχθεί και ότι το Συμβούλιο δεν θα χρονοτριβήσει καθόλου για να εγκρίνει κυρώσει ατομικές ε, ή ένα εμπάργο όπλων την στιγμή που θα δούμε ότι η διαδικασία του πολιτικού διαλόγου εκτροχιάζεται ή χρησιμοποιείται για κολλησιεργία. Τέλος θα ήθελα να χαιρετήσω τους ε, βουλευτές που βοήθησαν να, να ξεμπλοκάρει η κατάσταση στην Μανάγουα τον Ιανουάριο. Έτσι υπάρχει πλέον ένα περιθώριο για αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι ένας διάλογος σοβαρός ε, που θα στοχεύσει αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουμε λάβει έξι προτάσει ψηφίσματος για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Ολοκληρώνει τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης σχετικό με τη Διεθνή Δικαιοδοσία γνωρίσει και εκτέλεση αποφάσεων σε καμικέ διαφορές και διαφορές γονική μέρημνα και διεθνή απεγωγή παιδιών. Η συγγήτρια, η κυρία Πιτέρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πριν από ένα έτος ε, λάβαμε μία απόφαση για ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, ε, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε οικογενειακές διαφορές και για την διεθνή απαγωγή παιδιών. Το Συμβουλίο τελικά κατέληξε σε ένα μακρό έγγραφο. Το Κοινοβούλιο είχε υποστηρίξει την προηγούμενη έκθεση του κ. Βεύκα με μεγάλη πλειοψηφία και επισημάνομαι κάποιους τομείς σημαντικούς για εμάς. Παραδείγματος χάρη να ακουστεί το παιδί. Η χρήση διατησίας σε οικογενειακά ζητήματα. Χαιρόμαστε για το ότι έχουν περιληφθεί όλα αυτά στο τελικό κείμενο και είναι σημαντικό σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις όταν ένα δικαστήριο αποφασίζει ότι το παιδί θα πρέπει να πάει σε ανάδοχη οικογένεια Ε, πάλι το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα πρέπει να πάει σε αναδοχή οικογένεια ή με τους συγγενείς ή, οπουδήποτε αλλού, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίω και το πολιτιστικό υποβαθρό του παιδιού. Μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των αρχών μας θα επιτρέπει στα δικαστήρια να αποφασίζουν προς το συμφέρον ε, του παιδιού, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι ένα παιδί μια χι εθνικότητα θα πρέπει αυτομάτως να πηγαίνει στην οικογένεια της ίδιας εθνικότητας. Συγκεκριμένοι κανόνες ε, βεβαίως ε, θα ήταν χρήσιμοι, αλλά τα δικαστήρια, τα αρμόδια, θα πρέπει να είναι τα δικαστήρια της χώρας μόνιμης κατοικίας του παιδιού εάν συμφωνούν και οι δύο γονεί μπορεί να επιλεγεί διαφορετικό δικαστήριο ή το δικαστήριο το ίδιο μπορεί να αποφασίσει ότι θα πρέπει να κρίνει ένα διαφορετικό δικαστήριο προς το συμφέρον του παιδιού. Επίσης, όταν ένα παιδί επιστρέφεται μετά από απαγωγή από τους γονείς του, το ε, δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή του στην οικογένεια γιατί έτσι παραβιάζεται η αρχή του συμφέροντος του παιδιού ειδικά σε περιπτώσεις ε, συναισθηματικής ή σεξουαλικής ε, κακοποίησης του παιδιού. Επίσης, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, η ε, διαδικασία αυτή εξεκβάτουρ έχει καταργηθεί που δηλαδή την εκτέλεση της απόφασης δικαστηρίου άλλης χώρας. Τώρα τα κράτη-μέλη συνεργάζονται και το κείμενο αυτού του εγγράφου έχει λάβει υπόψη τις ε, διάφορες ε, καταστάσεις. Ε, μιλάμε για περίπλοκους τομείς της ζωής όπου σπανιότατα μπορεί να ληφθεί μια απόφαση που θα είναι άσπρη ή μαύρη. Το δικαστήριο λοιπόν πρέπει να καθοδηγείται από την αρχή του συμφέροντος του παιδιού. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την έκθεση την οποία παρουσιάζω εξ ονόματος κυρίας Βιέφκα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α είναι κλειδί για διασυνοριακά νομικά θέματα ε, σε γαμικές διαφορές και προστασία του παιδιού. Έχουμε προτείνει την διατύπωση αυτού του κανονισμού με στόχο να ε, προστατεύσουμε τα παιδιά σε διασυνοριακές ε, καταστάσεις, να μην καταλήγουν όμοιροι μακροσκελών διαδικασιών και έχουμε δει επίση ε, και το κόστος αυτών των διαδικασιών. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά θα πρέπει να καλύπτονται ε, ε, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη την οικογενειακή κατάσταση των γονέων. Τον Δεκέμβριο Φέτο οι Υπουργοί μετά από δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων συμφώνησαν για νέους κανόνες που θα παρέχουν καλύτερη προστασία των παιδιών και θα διευκολύνουν τις ε, διαδικασίες για τους γονείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας για αυτή την πρόταση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ε, τον, εισηγητή κ. Τσίφκα, για την εξαιρετική συνεργασία και την ε, επίσφαση της δεύτερης της ε, γνωμοδότησης. Θα δείτε ότι πολλά από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη γνωμοδότηση περιλαμβάνονται ε, στο συμβαστικό κείμενο. Από την άλλη πλευρά, το κείμενο δεν περιλαμβάνει όλα όσα ζητήσατε. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτοί οι κανόνες συμφωνήθηκαν με ομοφωνία. Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες και το κείμενο περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, ε, έχουμε καταργήσει τις ενδιάμεσες διαδικασίες για την διασυνοριακή επιβολή όλων των αποφάσεων, την ε, λεγόμενη exequatur. Ε, νέοι κανόνες για την επιβολή των αποφάσεων θα παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Στην διαδικασία επιστροφής του παιδιού χαίρομαι που θα υπάρχουν ε, βραχύτερες προθεσμίες για τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας αυτής. Το κείμενο ενισχύει τα δικαιώματα του παιδιού, διασφαλίζοντας ότι η προοπτική του παιδιού, ε, με μόνο μερικές εξαιρέσεις, ε, τη χάνει ακρόαση στις διαδικασίες. Η αμοιβαία αναγνώριση των πρακτικών των κρατών μελών θα αποφύγει την άρνηση ε, σε στάδιο αναγνώρισης ή επιβολής, επιτρέποντας μια πραγματική κυκλοφορία των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιπρόσθετα, ο συμβιβασμό θα παρέχει σαφέστερους κανόνες για την τοποθέτηση του παιδιού σε ένα άλλο κρατός μέλος ε, θεσπίζοντας αυτόνομη διαδικασία ε, συνένεσης και συγκατάθεσης όλων των ειδών τοποθέτησης. Οι κανόνες επίσης διασφαλίζουν μια πιο αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στις ιατρικές αρχές που θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στο να στηρίζουν τα δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές στο να εφαρμόσουν τους κανονισμούς. Προσβλέπω στις απόψεις σας και ε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει μεγάλη στήριξη για αυτό τον κανονισμό από το ε, Κοινοβούλιο αύριο στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοράτσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, συντονίστρια για τα παιδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζω τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 καθώς μας δίνει νέα μέσα για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση διασυνοριακών αποφάσεων για την ε, επιμέλεια και την απαγωγή παιδιών. Διευκολύνει την αποτελεσματικότητα των δικαστικών διαδικασιών. Παραδείγματο χάρη, όταν ένα ζευγάρι χωρίζει και ο ένας γονιός επιστρέφει στην χώρα πρόέλευσή του με το παιδί, χωρίς τον άλλον γονέα, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής του παιδιού. Αυτός ο κανονισμό επηρεάζει την καθημερινή ζωή πολλών οικογενειών και παιδιών. Και η διεθνής απαγωγή παιδιών έχει πολύ ε, σημαντικές συνέπειες για το παιδί. Όσο περισσότερο ε, διαρκεί, τόσο μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στη ζωή του παιδιού. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος. Γι' αυτό καλωσορίζω ιδιαίτερο το εξή ότι υπάρχουν ξεκάθαρα χρονικά όρια και για τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου και για την επιβολή τους περιορισμός στον αριθμό των εφέσεων που κατά κανόνα καθυστερούν τις αποφάσεις επιστροφής και υποχρέωση του δικαστηρίου να ακούσει και να λάβει υπόψη τις απόψεις των παιδιών σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να διατηρηθεί η αρχή του συμφέροντος του παιδιού. Και επίσης αναγνωρίζει το ότι το παιδί έχει δικαιώματα. Λυπούμε όμως για το ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφώνησαν σε κοινέ προδιαγραφές όσον αφορά τις ακροάσεις. Για να διασφαλιστεί, ε, να διασφαλιστεί ότι θα ακούει τη φωνή του παιδιού ε, δεν αρκεί και καμιά φορά μπορεί να επιβαρύνει το παιδί εάν δεν υπάρχουν κάποιες οικονομικές δικλείδες. Και ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των παιδιών που ασχολούμαι με πολλές τέτοιες περιπτώσεις ε, γονεϊκής απαγωγής έχω δει πως ε, συχνά αυτές οι διαδικασίες είναι τραυματικές για τα παιδιά. Οπότε ζητώ από εσάς ε, και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν κάποιες κοινέ προδιαγραφές και να δουν τις βέλτιστες πρακτικές για την διασφάλιση των παιδιών δεν πρέπει να υπάρχει διπλή θυματοποίηση του παιδιού και να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Επίσης χαίρομαι για το ότι μπαίνει εδώ και η διαιτησία. Συχνά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναζητηθούν μόνιμες λύσεις. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να προωθήσουμε την εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ των γονέων και των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε αυτές τις διαμάχες και Με αυτόν τον τρόπο θα επιληθούν γρηγορότερα οι διαφορές έτσι ώστε να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του παιδιού να βλέπει και τους δυο γονείς. Σας ευχαριστώ Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση των ε, παιδιών ε, σε διεθνείς γάμους ε, που διαλύονται γίνεται ακόμη πιο δύσκολη γιατί υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, ε, πολιτιστικές και νομικά συστήματα. Γι' αυτό είναι σωστό το ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση σε αυτόν τον ε, τομέα και χαίρομαι για το ότι έγιναν δεκτές ε, κάποιες προτάσεις που είχα κάνει στην έκθεσή μου ως διαμεσολαβήτρια του Κοινοβουλίου για τις διεθνείς απαγωγές γιατί αυτές είχαν προκύψει από την εμπειρία και την τριβή με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Γι' αυτό είναι θετικό το ότι οι διασυνοριακές αυτές ε, διαδικασίες επιταχύνονται. Υπάρχουν ξεκάθαρες διορίες ότι υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στην ε, διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το θετικό το οποίο χαιρετίζω. Και αυτό ήταν ένας λόγος για τον οποίο εμείς οι σοσιαλδημοκράτε, είπαμε ναι, είμαστε υπέρ μιας πιο γρήγορη διαδικασίας γιατί θέλουμε οι πολίτες να διευκολυνθούν το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό χάρηκα για το ότι στην ε, περίπτωση αυτή το Συμβούλιο πήγε πολύ παραπέρα από τις προηγούμενες περιπτώσεις που ήταν πολύ επιφυλακτικό. και βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει ακόμα να τα δούμε, τα οποία δεν είναι εντελώς ικανοποιητικά. Γιατί ισχύει αυτό μόνο για ε, παντρεμένα ζευγάρια και για όχι ε, για σύμφωνα συμβίωσης, γιατί υπάρχει δηλαδή αυτή η διάκριση εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ. Έχουμε αυτή την ε, παλαιού τύπου αντίληψη που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην ε, πραγματικότητα και είναι εδώ πέρα μια χαμένη ευκαιρία αυτή η υπόθεση. Ε, όπως επίσης και το ότι δεν έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές για την ακρόαση των παιδιών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ οι διαφορές, καμικές διαφορές ε, είναι δραματικές για τα παιδιά τα οποία είναι πάντα θύματα αυτών των διαφορών και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε πάντα το παιδί. Ε, αυτό που είναι δύσκολο είναι ότι μπορεί να πρέπει να προσφέρεις προστασία σε παιδί σε μια διαφορετική χώρα από την χώρα ε, καταγωγής του παιδιού το τελευταίο ψήφισμά μας ευστήσαμε την προσοχή σας στις καδαλώδεις πρακτικές ε, του γερμανικού Jugendamt όπου οι γερμανικές αρχές δεν επιτρέπουν στα παιδιά που ζουν στη Γερμανία να είναι σε επαφή με τους γονείς τους ε, ή ε, στη γλώσσα των γονιών του παιδιού. Το παιδί θα πρέπει να επιτρέπεται να διατηρήσει την πολιτιστική του ταυτότητα ε, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. Τώρα, αυτό που προτείνει η πολωνική κυβέρνηση είναι μια διαδικασία όπου με ταχύτητα και ευκολία μπορεί κανείς να ε, εντοπίσει συγγενείς του παιδιού που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη μέρημνά του. Ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις καναλαδόρες πρακτικές στην Γερμανία. κύριε Σκουφεράτη. Κύριε Πίτροπε, συζητάμε και θα ψηφίσουμε την τροποποίηση ενό ε, κανονισμού που είναι πολύ σημαντικό, είτε γιατί καθορίζει ομοιόμορφου κανόνε ε, για το διαζύγιο και την ακύρωση του γάμου και γιατί ε, παρεμβαίνει σε διασυνορικές ε, περιπτώσεις για τις γονικές ευθύνες συμπληρωματικά, ε, μάλλον συνολικά το κείμενο του Συμβουλίου θεωρείται ικανοποιητικό. Συμφωνούμε με τις περισσότερες τροποποιήσεις. Πιστεύουμε ότι είναι θετικό ότι το θέμα που αφορά την απαγωγή των παιδιών να είναι αντικείμενο καλύτερου συντονισμού στις κεντρικές ε, αρχές. Πιστεύουμε ότι είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί και η διαμεσολάβηση όπου είναι δυνατόν. Όμως είναι εντελώ απαράδεκτο να γίνεται όπως σήμερα, ε, να υπάρχει απόκληση μεταξύ των δικαιωμάτων ε, των πολιτών μελών. Ε, τα ίδια δικαιώματα δεν εφαρμόζονται στους συζύγους με την ίδια έννοια ή με όποιον έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και επομένως δεν θα μπορέσουν να υποφεληθούν καθόλου από τη δικαστική συνεργασία σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή από το κύριο νομοθέτημα της Ένωσης ε, που ρυθμίζει τα διαζύγια και την ακύρωση του γάμου ε, όπως και τις διαφορές γονικής μέρημνας. Ε, τελικά λέμε ότι υπάρχουν πολίτες κατηγορίας Α και πολίτες κατηγορίας Β με κατώτερα δικαιώματα. Αυτό είναι εντελώ απαράδεκτο. Έχουμε παρουσιάσει διάφορε τροπολογίε προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή, όμω δεν θεωρήθηκαν παραδεκτέ. Πιστεύουμε ότι και αυτό είναι μεγάλο λάθο και είναι λάθο το να μην καλύπτουν όλους τους πολίτες τα ίδια δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βόρτ. Uh, thank you, President. This ευχαριστώ. Η πρώτη και κύρια ευθύνη αυτού του κοινοβουλίου είναι να προστατεύει του πολίτε και ειδικά του πιο ευάλωτου. Και αυτή είναι τα παιδιά. Έχουμε συγκλονιστικέ περιπτώσει όπου αμφισβητείται η επιμέλεια των παιδιών, ειδικά σε περιπτώσει ε, διεθνού απαγωγή. Σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα νομικά μέσα, χωρί γκρίζε ζώνε και παραθυράκια. Καλωσορίζω πολλά σημεία αυτή τη πρόταση, ειδικά την υποχρεωτική ακρόαση του παιδιού ως συνειδητής ε, της ε, ομάδας για τα δικαιώματα του παιδιού σε αυτό το κοινοβούλιο θεωρώ ότι οι φωνές των παιδιών πρέπει να ακούγονται σε ζητήματα που τα αφορούν. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος. Οι οικογένειες ε, σημαίνουν πολλά πράγματα και θα πρέπει να περιληφθούν εδώ πέρα και τα σύμφωνα συμβίωση. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει ότι αντιλαμβάνεται τι πολλέ μορφέ μια οικογένεια. Καθώ αν δεν το κάνουμε, θα έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα για τα παιδιά. Όπω φαίνεται από πολλέ περιπτώσει διεθνού απογωγή. Σα ευχαριστώ. Κινίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα πάνω από 16 εκατομμύρια οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούνται από γονεί που έχουν διαφορετική εθνικότητα και αυτό αποτελεί συνέπεια τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Όμω χρειάζεται ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να ρυθμίζονται οι οικογενειακές διαφορέ και να προστατεύονται τα παιδιά. Σύμφωνα με την ε, πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν έχουμε περίπου 1.800 ε, περιπτώσεις ε, διεθνούς απαγωγής παιδιών, δηλαδή όπου και δύο ή τα διεκδικούν. Η διατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α έρχεται για να επικαιροποιήσει ε, αυτό το τομέα και εισάγει θετικές καινοτομίες, κυρίως επιβάλλοντας στις δικοστικές αρχές ε, την υποχρέωση της ακρόασης του ανηλίκου ακόμη ε, και αν η διάταξη θα μπορούσε να έχει ενταχθεί με μία παραπομπή ε, στους τρόπους της ακραίωσης ε, και σε διάφορους τρόπους προστασίας του παιδιού από τα τραύματα. Θα πρέπει να προωθηθεί μια οικογενειακή διαμεσολάβηση για να επιληθούν οι διαμάχες μεταξύ των γονιών, κυρίως προς το συμφέρον του παιδιού, γιατί τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να προστατεύονται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο ΚΑΤΣΔΙ. Ο κύριος Ποσπισίλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω αυτή την αλλαγή στον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Εγώ ήμουν υπουργό δικαιοσύνη και θυμάμαι ότι τα δικαστήρια εφάρμοζαν διαφορετικές διαδικασίες στα διάφορα κράτη-μέλη σε ε, περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών. Καλωσορίζω λοιπόν ε, αυτή τη διευκρίνηση στις Βρυξέλλες 2α. Ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθει πιο κοντά η πρακτική στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, καλωσορίζουμε τις προθεσμίες γιατί στο παρελθόν είδαμε πάρα πολλές καθυστερήσεις σε διάφορες υποθέσεις που αφορούσαν παιδιά. Αυτό αποτελεί μια καλή πρόοδο. Επίσης, καλωσορίζω το σημείο για την υποχρεωτική ακρόαση του παιδιού. Όλα αυτά ωφελούν τα παιδιά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ε, μεικτά ε, ζευγάρια και δυστυχώ έχουμε διεθνεί περιπτώσει περιπτώσεις παιδιών. Ευχαριστώ. Κύριος Λόπε Αγγιλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι ή δεν είναι γιγάντιο βήμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά έχει νομοθετική ικανότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι φορά το οικογενεικό δίκαιο από τη στιγμή που ψηφίστηκε η συνθήκη τη Λισαβόνα και για το θέμα τη ακύρωση του γάμου, του διαζυγίου ή των ε, γονικών υποχρεώσεων σε διασυνορικέ υποθέσει. Φυσικά και είναι. Αλλά αυτό το γιγάντιο βήμα έχει και περιορισμού στην ομοφωνία συμβουλίου και ε, την ε, διαδικασία διαβούλευση που ακολουθείται στο Κοινοβούλιο. Και παρόλα αυτά θεωρούμε ότι γίνεται ένα θετικό βήμα για την ε, κατάργηση του εξεκβάτουρ, ε, για την αποσαφήνιση των κανόνων ε, σε σχέση με την απαγωγή των παιδιών και την αμοιβαία αναγνώριση των διασυνοριακών δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, είναι ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε και τι εκρεμεί. Η αναγνώριση των διάφορων μορφών οικογένεια, τα de facto γευγάρια, τα ζευγάρια των ομοφύλων, ομοφυλοφίλων. Στην περίπτωση τη Ισπανία να αναγνωρίζονται αυτά και να υπενθυμίσω πόσο σημαντική είναι ε, η ενίσχυση νομοθετική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και φυσικά αυτά θα αποφασιστούν και στις ευρωεκλογές 26 Μαΐου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του κανονισμού 2201-2003 πραγματικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς καλύπτει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων του οικογενειακού δικαίου διότι όπως γνωρίζουμε έχουμε διεθνείς γάμους και φυσικά πολλές φορές προκύπτουν διαζύγια ακυρώσεις γάμων και μάλιστα μεγάλες διαφορές γύρω από την γονική μέρημνα των παιδιών όπως επίσης και για τις υποχρεώσεις των γονέων όπως είναι η υποχρέωση διατροφής. η διαδικασία επιστροφής των παιδιών είναι μια σημαντική διαδικασία καθώς έχουμε πολλές φορές απαγωγή του τέκνου πολλές φορές έχουμε και τοποθέτηση του παιδιού σε ένα άλλο κράτος δηλαδή δίδεται σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ένα ίδρυμα και στην επιτροπή αναφορών είχαμε πολλές καταγγελίες για την διακριτική μεταχείριση που ε, κάνει το περίφημο jugendamt στη γερμανία εις βάρος των ευρωπαίων πολιτών που δεν είναι γερμανοί. θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά που συζητούμε είναι ενδιαφέροντα είναι πολύ σημαντικά πρέπει να λυθεί το θέμα της κήρυξης της εκτελεστότητας της απόφασης και φυσικά να υπάρχει η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων. πολύ δε περισσότερο να περιοριστεί και η διαδικασία με τα πολλά ένδικα μέσα. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Μαριά. συνάδελφοι. Όπως έχει ήδη με τη βελτιωμένη κινητικότητα έχουμε και τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αξίζει να τα ε, παρακολουθούμε και να αντιδρούμε. Σε αυτή τη περίπτωση με νέα νομοθεσία λόγω πολλαπλών γάμων ανάμεσα σε ε, διαφορετικές εθνικότητες ε, προκύπτουν περισσότερες ε, διασυνοριακές δικαστικές διαφορές. Από την πράξη ξέρουμε ότι οι διαδικασίες είναι μακρό ε, και οι ερμηνείες των δικαστηρίων διαφέρουν. Αυτό έχει αντίκτυπο στα παιδιά που ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Η αυτόματη επιβολή της ε, δικαστικής απόφασης και η συνεργασία των αρχών των κρατών μελών που λαμβάνουν τις δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να συμβάλλουν προς βελτίωση των διαδικασιών. Το συμφέρον του παιδιού θα είναι η προτεραιότητα και αυτό ε, το συμφέρον είναι να μην υπάρχουν διαζύγια. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που περίχε πάρα πολλά έγκυρα σημεία. Η ψηφοφορία σας αύριο θα ε, οδηγήσει στην επιτυχή, ε, ε στο επιτυχή κλείσιμο των πραγματεύσεων υπό αυτή την Προεδρία, έτσι ώστε να εφαρμοστούν νέοι κανόνες και να βοηθήσουμε ε, οικογένειες σε αυτές τις καταστάσεις και να προστατεύσουμε κυρίως τα παιδιά. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο και όσους πήραν το λόγο για τη συνεισφορά τους. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμήνεις. Ευχαριστούμε και εμείς. Η επόμενη σύνοδος θα λάβει χώρα αύριο στις 14 Μαρτίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η μερεσία διάταξη έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ολοκλήρωση της συνεδρίασης.